Bien, chacun a pu gagner sa place. Καθίστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας καλωσορίζω από βάθους καρδίας σε αυτήν την ε, Διακοινοβουλευτική Επιτροπή που είναι αφιερωμένη στα ζητήματα των προπολογισμών. Χαιρετίζω μεταξύ μας και την παρουσία της κυρίας Κρυσταλίνα Γεώργεβα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνη για τον προπολογισμό και για τους ανθρώπινους πόρους. Πριν από λίγο καιρό ακόμα ερχόμουν εδώ στις Βρυξέλλες και συμμετείχα σε τέτοιες συναντήσεις ως εθνικός βουλευτής. Τότε ήμουνα στην Επιτροπή Οικονομικών της Γαλλικής Γερουσίας. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σας υπό άλλη ιδιότητα, υπό την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή και Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Άλλαξα όργανο, άλλαξα σώμα, η αποστολή μου όμως παραμένει ίδια. Πρέπει να φροντίσουμε η διακυβέρνηση να γίνεται αποτελεσματικά και με θάρρος προκειμένου να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους οι συμπολίτες μας. Και είμαι πεπισμένος ότι μέσα στην παγκοσμιοποίηση, μέσα σε ένα κόσμο με τεράστιες αλλαγές, οι χώρες μας δεν θα τα βγάλουν πέρα χωρίς την Ευρώπη. Και συγχρόνως η Ευρώπη δεν θα ολοκληρωθεί χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις όλων των χωρών μελών και το συντονισμό των δράσεών τους. Δηλαδή το καθήκον μας είναι να υπάρξει συνεργασία, να ακούσουμε μεν τους δε τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τις επιθυμίες των συντονιστών της Επιτροπής Προπολογισμών θα ήθελα να προσέξετε εδώ πέρα μια δυσλειτουργία που έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές πιστώσεις. Φυσικά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην απόφαση για υποχρεώσεις πιστώσεων και, τον, ε, και τις πληρωμές που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και πολλά χρόνια οι λογαριασμοί συσσωρεύονται στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν γιατί δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Και έτσι καταλήγουμε σε μια χιονοστιβάδα που όλο γίνεται μεγαλύτερη. Στις 31 Δεκεμβρίου είχαμε 23 δισεκατομμύρια ευρώ απλήρωτους λογαριασμούς. 5 δισεκατομμύρια από το 2010, 11 δισεκατομμύρια στα τέλη του 2011, 16 στα τέλη του 2012 και σήμερα στα τέλη του 2014 δηλαδή είμαστε στα 25 δισεκατομμύρια. Συνεπώς, κυρία Αντιπρόεδρε, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν φτάσει σε μένα. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με ένα συνεχώς αυξανόμενο χρέος. Το έλλειμμα επίσης αυξάνει κάθε χρόνο και καταλήγει να είναι διαρθρωτικό. Βέβαια οι νομικοί θα σας εξηγήσουν ότι οι λογαριασμοί δεν είναι χρέη έτσι όπως αυτοί στις συνθήκες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν φορείς οι οποίοι περιμένουν να πληρωθούν για προγράμματα τα οποία έχουν αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς υπάρχει ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια σκοτεινή εικόνα της Ευρώπης Χρειάζεται συνεπώς να διορθωθεί η κατάσταση αυτή όσον αφορά τον προϋπολογισμό και να μην καταλήξουμε να είμαστε κακοί πληρωτές. Αυτό πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς ε, τεχνοκρατικές ε, αντιμετωπίσεις. Έχουμε εδώ πέρα ε, εκπροσώπους των τοπικών αρχών και θα ακούσουμε τις δικές τους μαρτυρίες για να καταλάβουμε καλύτερα. Χρειάζεται να είμαστε πιο ξεκάθαροι και να έχουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Πώς φτάσαμε πρώτα απ' όλα εδώ, πώς μας ξέφυγε έτσι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως όλοι μαζί μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι λάθη υπάρχουν σε διάφορες πλευρές. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο μέρος ευθύνης έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις των χωρών ε, μελών που εκπροσωπούνται από τους Υπουργούς Οικονομικών οι οποίοι συνεδριάζουν στο Συμβούλιο. Βέβαια, στον πρώτο τέτοιο κύκλο δημοσιονομικό θυμάμαι ότι δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο να μιλήσω με 28 υπουργού προπολογισμών. Μόνο ένα Ιταλό ήρθε να συναντηθεί με του 28 ε, ε, ευρωβουλευτέ τότε που ήταν στην διαπραγματευτική ομάδα. Έπειτα υπάρχουν υπηρεσίε, υπρέψει κτλ. οι οποίοι είναι περισσότερο διακοσμητικοί γιατί δεν μπορούν να έχουν ε, θέση. Και όλα αυτά μέσα βέβαια σε μια λογική βράχη πρόθεσμη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσε δυσκολίε των χωρών μελών, να ισορροπήσουν του δικού του εθνικού λογαριασμού. Και αυτό έρχεται σε αντίφαση βέβαια με τι δεσμεύσει που είχαμε αναλάβει κατά το παρελθόν. Θυμάμαι την ε, καγκελάριο Μέρκελ και τον πρόεδρο Ολάντ το, το φθινόπωρο του 2013 που είχαν ανακοινώσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και τον Νοέμβριο 2014 είπαν ότι δεν υπήρχε επαρκής προχρηματοδότηση από πλευρά στην Ευρώπη και το Δεκέμβριο οι κυβερνήσεις τους αρνήθηκαν να τιμήσουν τις υποχρώσεις που είχαν αναλάβει προηγουμένω. Συνεπώς πρέπει ο λόγος που δίνουμε να τηρείται. Αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς που είσαστε στα εθνικά κοινοβούλια, μιλήστε στους υπουργούς σας οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους και βάζουν πολλούς φορείς σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είτε πρόκειται για τις τοπικές αρχές, για τις περιφερειακές, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για εργαστήρια ερευνητικά, για μη κυβερνητικέ ανθρωπιστικές οργανώσεις κλπ. Αυτή η κατάσταση πλήττει την ίδια την ανάπτυξη για την απασχόληση. Κάτω από αυτέ τι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει χωρίς να έχει καθαρό τοπίο. Το σύστημα είναι μάλιστα τόσο αδιάφωνο και περίπλοκο που δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις για τα οικονομικά. Χωρίς να μπορούν λοιπόν να έχουν ορατότητα, δεν μπορούν να δώσουν κατεύθυνση, να προλάβουν. Παίρνουν από μία δημοσιονομική γραμμή για να βάλουν χρήματα σε μια άλλη γραμμή του προπολογισμού κλπ. Ε, αυτό σχεδιάσουμε. Καθυστερούμε τις προθεσμίες. Ε, γι' αυτό πολλαπλασιάζουμε τις διοικητικές ε, διαδικασίες και βρίσκουμε προσχήματα. Έχουμε να κάνουμε με μια Ευρώπη γραφειοκρατική, κατακαιρματισμένη. Πρέπει όμως να αλλάξει. Εσείς, κύριε Πίτροπε Γεωργιεβά, που αναλάβατε πέρυσι τα καθήκοντά σας όπως και εγώ, δεσμευθήκατε με τι διαπραγματεύσει του προπολογισμού του 2014 να βάλετε τάξη στα βιβλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνετε του λογαριασμού να αποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα και να μπορούν να ελεγχθούν από την Επιτροπή των Προπολογισμών. Και όταν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι υπεύθυνοι για τον προπολογισμό εξετάζουν όλα αυτά τα θέματα, καταλήγουν στο ότι πρέπει οι λογαριασμοί να πληρωθούν. Χωρί να ε, είμαι προκλητικό ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αναλύσει την οικονομική κατάσταση των χωρών μελών να συμπεριλάβει παρακαλώ εκτός από το έλλειμμα και το χρέος το κομμάτι των χωρών μελών που αντιστοιχεί σε αυτούς τους απλήρωτους λογαριασμούς. Γιατί οι απλήρωτοι αυτοί λογαριασμοί που συσσωρεύονται στις Βρυξέλλες είναι χρέος των χωρών μας. Το Κοινοβούλιο φταίει και αυτό, αλλά έχει και κάποια δικαιολογία. Και αυτή είναι ότι η η διαδικασία του προπολογισμού έτσι κι αλλιώς είναι ανάπηρη ιστορικά, γιατί συνήθως τα κοινοβούλια αποφασίζουν και για τους φόρους, για τέσσερα, ενώ το δικό μας το σώμα δεν συλλέγει φόρους, δεν έχει λόγο στους πόρους, έχει μόνο ένα όπλο στη διάθεσή του και αυτή είναι η απόφαση για τις υποχρεώσεις δαπανών. Τα πράγματα μπορούν να αρχίσουν να αλλάξουν. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλού επίπεδου υπό τον Μάριο Μόντι για να ε, δώσει στην Ευρώπη πραγματικού ίδιου πόρου. Οι ίδιοι πόροι αυτοί θα ενισχύσουν την θεσμική αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την εικόνα του τη θεσμική και συγχρόνως, θα ανακουφιστούν οι προπολογισμοί των χωρών μελών, δικοί σα προπολογισμοί, γιατί θα μειωθούν οι συνεισφορέ οι εθνικέ στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε φιλόδοξοι, να είμαστε δημιουργικοί, αλλά να μην προσθέσουμε στους εθνικούς φόρους και το βάρος ενός επιπλέον ευρωπαϊκού φόρου. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, Ζητάω τη βοήθειά σα για να αξιολογήσουμε την πραγματικότητα των απλήρωτων λογαριασμών στι δικέ σα χώρε. Σα καλώ λοιπόν να ενώσετε τι δικέ σα προσπάθειε με τι δικέ μα για να ελέγξουμε τι δημόσιε δαπάνε και να βεβαιωθούμε ότι οι προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια πραγματική προστιθέμενη αξία και ότι συνεισφέρουν οι προσπάθειες αυτές πραγματικά να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Επίσης κάνω έκκληση και στην κοινή λογική. Έχουμε ένα κοινό χώρο. Πολλοί από εμάς μοιραζόμαστε ένα κοινό νόμισμα, κοινέ ε, συνήθειες και νοοτροπίες στον προπολογισμό αλλά ένας πραγματικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρειάζεται. Γιατί σήμερα έχουμε ένα, μια συσσόρυβη, μια πρόσθεση εθνικών προϋπολογισμών και όχι ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και αυτή είναι η δυναμία μας. Και γι' αυτό επήγει να υπάρξει πιο ομοιογενής παρουσίαση και αξιολόγηση των εθνικών λογαριασμών. Έχουμε φτάσει στο τέλος ενός κύκλου. Πρέπει να ακούσουμε τα μηνύματα που μας στέλνουν οι πολίτες μας και που μας στείλαν στις ευρωεκλογέ το Μάιο του 2014. Η Ευρώπη αποτελεί αντικείμενο αφιβολιών και επικρίσεων. Χρέος μας είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα το business as usual. Πρέπει να ξαναδούμε τις μεθόδους με τις οποίες εργαζόμαστε να γίνουν πιο κατανοητές οι πρακτικές που ακολουθούμε και αυτό για να βοηθήσουμε την Ευρώπη να σωθεί. Χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν δώσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Γιώργεβα, θα ήθελα να σας πω και δύο λόγια για το πώς θα προχωρήσουμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδριάσεώς μας θα έχουμε διερμηνία προς όλες τις γλώσσες πλην των Μαλτέζικων. Στις 12 και 4 θα πάψουμε να έχουμε μαλτέζικα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να περιορίσετε τον ε, χρόνο των παρεμβάσεών σας, δύο λεπτά το πολύ, για να μπορέσουν όσο γίνεται περισσότεροι να παρέμβουν. Έχετε κάρτες, speaking cards, στις θέσεις σας. Για να ζητήσετε το λόγο λοιπόν πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην κάρτα αυτή και να τη δώσετε σε έναν κλητήρα. Αυτό ισχύει για τους εθνικούς βουλευτές αλλά και για τους ευρωβουλευτές κατά τις παρεμβάσεις σας. Να ξέρετε ότι θα έχουμε δύο από το Εθνικά Κοινοβούλια και έναν Ευρωβουλευτή. Συνεπώς, κύριε Αντιπρόεδρε, υπεύθυνοι για τον προπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι, των Κοινοβουλίων, κύριε και κύριοι. Με μεγάλη χαρά λαμβάνω το λόγο ενώπιον των μελών των Επιτροπών Προπολογισμού. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Αρτιού για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τη γενική προβληματική στην ομιλία του και επίσης και στο έγγραφο εργασίας το οποίο έχει προετοιμαστεί ήδη πριν από τη συνεδρίασή μας. Είναι δύσκολη η χρονική στιγμή για την Ευρώπη. Παρά τις προσπάθειές μας εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε ακόμα για να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης που βαραίνει σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο νοικοκυριού. η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει πληγεί από την κρίση αυτή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πράξω θα ήταν να εστιάσω περισσότερο στο θέμα των πιστώσεων πληρωμών που ανέφερε και ο πρόεδρος Σαρτουή προηγουμένως αλλά θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην ευκαιρία μετα... μεταρρύθμισης που μπορεί να γίνει παρά την στενότητα του προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό να έχουμε ένα προπολογισμό που να εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα και να αναφερθώ στις προτεραιότητες της Κομισιόν σε αυτή την ενδιάμεση στιγμή που γίνεται η ενδιάμεση μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών προοπτικών και να σκεφτούμε και για τη συνέχεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Ξεκινάμε λοιπόν με τις πιστώσεις πληρωμών. Είναι φανερό ότι είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Αυτό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Πρέπει να πληρώσουμε τα οφειλόμενα. Αλλά ήμασταν κάπως απροετοίμαστοι για το τέλος της εποχής των παχαίων αγελάδων να το πω πιο σαφώς, για δεκαετίες ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έδινε περισσότερες πιστώσεις πληρωμών, ικανότητα δαπανών, από ό,τι χρειαζόταν να γίνουν πληρωμές. Κάθε χρόνο, λοιπόν, γινόταν αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν μια εσφαλμένη εντύπωση απεριόριστων πόρων. Γιατί τα κρατημέλη τα ίδια και η Κομισιόν είχαν δυσκολία να απορροφήσουν τους διαθέσιμους πόρους. Κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ έμεναν αδαπάνητα. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια κουλτούρα εύκολων δαπανών. Αυτό όμως έφτασε στο τέλος της όταν ξαφνικά οι πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν να ελείπουν και όταν η ζήτηση για αυτούς τους πόρους συγχρόνως άρχισε να αυξάνεται. Αυτό αντιμετωπίσαμε το 2010, 2011, 2012 ήδη τα κράτη-μέλη μας, τα οποία πλήγησαν από την κρίση, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον χρειάζονται για τα εθνικά τους σχέδια περισσότερο, ενώ συγχρόνως υπάρχει η τροπή προς τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές από το 2014, όπου τα χρήματα τα οποία διαθέσιμα για την περίοδο προγραμματισμού την τρέχουσα ήταν λιγότερα από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Το 2013 και το 2014 είδαμε να συσσωρεύονται οι απλήρωτοι λογαριασμοί και αγωνιζόμαστε να εξασφαλίσουμε την αποπληρωμή αυτών των λογαριασμών χωρίς να υπονομεύσουμε τα προγράμματα της νέας δημοσιονομικής περίοδου. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί στις διαπραγματεύσεις για τους νέους για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη ευκαμψία, μεγαλύτερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και πολύ ορθώς. Όταν πρέπει να διαχειριστούμε ένα λιτό προϋπολογισμό θα πρέπει να έχουμε μια πιο εύκαμπτη αντιμετώπιση από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή η ευκαμψία είναι αυτή η οποία μας διέσωσε, γιατί το 2014 βρεθήκαμε σε θέση να δανειστούμε ή εν να μετακομίσουμε πιστώσεις ε, για να τις χρησιμοποιήσουμε το 2014 από τα επόμενα έτη που ελπίζουμε θα υπάρχουν λιγότερα προβλήματα για τη χρηματοδότηση. Υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να μετακομίσουμε κονδύλια στο 2014 και έτσι μπορέσαμε να αναχαιτήσουμε την αύξηση της ισόρευση λογαριασμών. Ε, έχουμε καταλήξει λοιπόν σε 25 δισεκατομμύρια σε απλήρωτους λογαριασμούς σήμερα το 2015, αλλά είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να έχουμε ένα σχέδιο αποπληρωμής, ώστε η κατάσταση αυτή να διορθωθεί το 2015 και το 2016. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το σχέδιο για την πληρωμή αυτή των οφειλωμένων. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να επιτευχθεί μια βελτίωση στην ποιότητα των δεδομένων και στην συνεκτικότητα των δεδομένων, ώστε να κάνουμε καλύτερες προβλέψεις για τις ταπάνες μας, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων. Όταν δεν έχει κανείς περιορισμούς, όταν έχει δυνατότητα απλόχερα να πληρώνει κανείς γιατί έχει περισσότερα χρήματα από ό,τι χρειάζεται να πληρώσει, μπορεί κανείς να είναι χαλαρός στη διάρθρωση των προγραμμάτων του. Αλλά τώρα που υπάρχει στενό της προπολογισμού, είναι κεφαλαιώδης ικανότητα καλύτερου σχεδιασμού και καλύτερης υλοποίηση των ευρωπαϊκών σχεδίων. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ικανότητα πρόβλεψή μας και τη συνεκτικότητα των στοιχείων μας. Και επίση, όπω γνωρίζουμε πολύ καλά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο είναι πολύ δημοφιλές. Α, δεν πιστεύουμε τις προβλέψεις σας, ξανακάντε τις και ελάτε και βοηθήστε μας να κάνουμε εξοικονομήσεις. Αλλά τώρα φαίνεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε τόσο εύκολα εξοικονομήσεις. Δεύτερον, τα τελευταία χρόνια και ιδίω το 2014 έχουμε αναλάβει μια σειρά από μέτρα σε διάφορους τομείς ταπανών ώστε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν κάπως ad hoc τα μέτρα αυτά. Είχαν διαφορετική μορφή σε διάφορους τομείς. Εγώ ήμουν τότε επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας και εμείς προσκούσαμε πρώτοι σε μια έλλειψη πιστώσεων πληρωμών και ξέρω πολύ καλά πώς χρειάστηκε να τροποποιήσουμε τις ε, διαρθρώσεις των δαπανών μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτά τα μέτρα λοιπόν τώρα θεσμοποιούνται ώστε να είναι τμήμα της όλης διαδικασίας πληρωμών. Και τώρα, το 2016, τι πρέπει να γίνει στον προϋπολογισμό του 2016 για να βοηθηθεί η ομαλοποίηση της κατάστασης των πληρωμών που οφείλονται. Προφανώς θα αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα για τον δυνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Το σχέδιο πληρωμών να είναι κάτι που το υποστηρίζει όχι μόνο η Κομισιόν αλλά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο γιατί από αυτό εξαρτάται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε μια καλή εικόνα ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν οι μικρές επιχειρήσεις, οι, οι ερευνητές, οι μεμονωμένοι, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν ξέρουν καν κατά πόσο θα τους πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα οφειλόμενα ποσά. Μετά από δεκαετίες αξιοπιστίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποσκάψει και να διαβρώσει αυτή την αξιοπιστία και να μειώσει τη σημασία που έχει για την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και για την εμπιστοσύνη της οποίας χαίρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως έμπιστος εταίρος και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της. Έχω κάθε εμπιστοσύνη για το ότι εμείς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι στο τέλος του 2016 θα έχουμε πετύχει μια ουσιαστική βελτίωση σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Πιστεύω ότι εν καιρό θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε επιτυχώς αυτή την προσαρμογή από τις εποχές αυθονίας στις εποχές στενότητος του προϋπολογισμού. Πιστεύω επίσης ότι αυτό αποτελεί και μια ευκαιρία για μας όταν έχει κάνει στενότητα προπολογισμού, οπωσδήποτε θα πρέπει κανείς να εστιάσει στην προσθέμενη αξία αυτού του προπολογισμού <clears throat> και τους στόχους που εξυπηρετούνται, ώστε να εστιάσουμε επίση στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της χρήση του προπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ως αρμόδια για τον προπολογισμό, εγώ ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να εξασφαλίσω την σφυριλάτηση μιας κοινή θέση μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβουλίου, αλλά και κυρίως μεταξύ και των κρατών μελών, ώστε, θα, ώστε να έχουμε ένα προϋπολογισμό που να εστιάζει στα αποτελέσματα. Και αυτός να είναι ο κοινό παράγοντας, ο κοινό παρανομαστής στον αγώνα μας για ανάπτυξη και καλύτερη απασχόληση. Να δημιουργήσουμε ισοδίκαιες συνθήκες για όλους στην Ευρώπη, γιατί γνωρίζουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης η ανεργία είναι εξαιρετικά υψηλή, είναι δύσκολο να μειωθεί. Τα δύο τρίτα των κρατών μελών μας είδανε να αυξάνεται το ποσοστό των ενδεών για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απόλυτη υποχρέωση να εστιάσει τον προπολογισμό μας στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αντικτύπου που προκάλεσε η κρίση. Και δεν είναι κάτι το οποίο μας κατέλαβε εξαπίνης. Είδαμε τον προϋπολογισμό μας να δημιουργεί απασχόληση και ανάπτυξη. Υπάρχει μια αξιόπιστη μελέτη που καταδεικνύει ότι για τη Λετωνία η χρηματοδότηση με το Ταμείο Συνοχής οδήγησε σε 2,5% πρόσθετη ανάπτυξη, 8% για τη Λιθουανία, 1,7% για την Πολωνία. Αυτό βοήθησε αυτές τις οικονομίες βοηθάει όλη την Ευρώπη γιατί είμαστε αλληλοσυνδεδεμένες σε επίπεδο οικονομίας. Και τώρα το σχέδιο Juncker θέλει να κάνει κάτι πολύ σημαντικό, να χρησιμοποιήσει ως βάση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ώστε με μόχλευση να μπορέσει να υπάρξει κινητοποίηση της υπνότουσας ρευστότητος στο τραπεζικό μας σύστημα και να μπορέσει να κατευθυνθεί προς στρατηγικές επενδύσεις να μπορέσουμε να έχουμε εξ αυτών των ποσών 75 δισεκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ελπίσουμε. Εάν εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο Juncker θα δημιουργήσει 2,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Μια τέτοια αντιμετώπιση θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να την επιβάλλουμε στον εαυτό μας κάθε μέρα, όχι πόσα πόσα δαπανούμε, αλλά τι θα αποκομίσουμε ως Ευρωπαίοι από αυτή τη χρηματοδότηση, αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη που επομιζόμαστε για τη σωστή χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων και τη σωστή λογιστική απεικόνηση των αποτελεσμάτων. Και εδώ είναι ιδιαίτερα προσφυλωμένη η νέα Κομισιόν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και μια ομάδα εργασίας διαθυσμικού επίπεδου για να παρακολουθούμε την απόδοση των μέτρων αυτών με συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά και του Συμβουλίου και επίσης στην καθημερινή μας εργασία. Θέλουμε να φέρουμε από κοινού την Κομισιόν και τα κρατημέλη για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη λογοδοσία. Κλείνοντας, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ενδιάμεση αναθεώρηση. Παραδοσιακά, τις εποχές της αυθονίας δεν ήταν τόσο σημαντική αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση. Αλλά τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα και το Κοινοβούλιο επέμεινε να πάρουμε πολύ στα σοβαρά αυτή τη μεταρρύθμιση και την ενδιάμεση αναθεώρηση. Θα πρέπει να δούμε τώρα πώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες, τι θα κάνουμε για να ανταποκριθούμε σε αυτές. Όταν υπήρχαν εποχές αυθονίας δεν υπήρχαν αρνητικές προτεραιότητες, είχαμε αρκετά για όλα. Τώρα πρέπει να σταθούμε πολύ πιο σόφρονες σε σχέση με τη στοχοθεσία και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Έχουμε 10 προτεραιότητε ω Νέα Κομισιόν. Προσπαθούμε να αναρμονίσουμε τον προπολογισμό με αυτέ τι προτεραιότητε. Θέλουμε όμω συγχρόνω να προσαρμόσουμε τον προπολογισμό στην αλλαγή των προτεραιοτήτων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 7 χρόνια τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι αλλαγέ. Στην ενδιάμεση λοιπόν αναθεώρηση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και μερικά ουσιαστικά ερωτήματα ουσίας και να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Μία από αυτές τις βασικές προβληματικές θα προέλθει από την ομάδα Μόντι για τους ίδιους πόρους και είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Ποιε πρέπει να είναι οι πηγέ του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ πρέπει να χρηματοδοτείται, πού είναι, ε, που είναι οι ελλείψει του τωρινού συστήματο, πώ πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μέσα από αυτή τη συζήτηση για του ίδιου πόρου, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή, αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Κάθε, σε κάθε βήμα χρειαζόμαστε την ομοφωνία. Θα πρέπει και τα 28 κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο να συνέσουν σε αυτή τη μεταρρύθμιση που είναι απαρέγκλητη. Και το τελευταίο σημείο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας να καθορίσουμε σαφώς πού βρίσκεται η προσθέμενη αξία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ποιες είναι οι παράμετροι μέσα στους οποίου θα πρέπει να επιτύχουμε τους κοινού μας στόχους, την Ενεργειακή Ένωση, την ψηφιακή ενιαία αγορά είναι σημαντικά θέματα για την επόμενη περίοδο προπολογισμού. Τι χρονικό διάστημα θα πρέπει να καλύπτει, λειτουργούμε τώρα με επταετή περίοδου, ίσω όμω χρειάζεται ένα πιο μικρό χρονικό διάστημα. Και πάνω απ' όλα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να έχουμε μεγαλύτερη ενότητα, μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος είναι ο στόχος της ύπαρξής της. Ο προπολογισμό είναι απλώ μια υποστήριξη, ένα εργαλείο υποστήριξη για την επίτευξη των κοινών μα στόχων. Είναι ένα μέσο και όχι ένα αυτοσκοπό. Εδώ ελπίζω ότι εσεί ω κοινοβουλευτικοί, ευρωπαίοι και εθνικοί θα μπορέσετε να παίξετε ένα κεφαλαιόδη ρόλο. Και από την πλευρά της Κομισιόν λοιπόν, ο στόχος μας είναι εργασία, εργασία και περισσότερη εργασία. Είναι υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε για αυτό τον κοινό στόχο και οι υπάλληλοι μου και εγώ θα το πράξουμε. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ κυρία μου. Είναι στενές οι σχέσεις μεταξύ ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον ε, κύριο Αντρέη Γαλαζεύσκη, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πολωνικής Βουλής. Εγώ να μιλήσω πολωνικά αφού σας ευχαριστήσω πρώτα κύριε Πρόεδρε και για όλους καλύτερα και για μένα καλύτερα και πιο εύκολα. για την κρίση πληρωμών. Πρώτα όμως να μιλήσω εγώ για μια άλλη κρίση, την κρίση εμπιστοσύνης Νομίζω ότι είναι αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης που εξακολουθεί να υπάρχει. Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα της έλλειψης αυτής της εμπιστοσύνης. Βλέπουμε την ενίσχυση των διαφόρων λαϊκιστικών κινήσεων, ακραίων λαϊκιστικών κινήσεων. Το πρόβλημα είναι οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και η υποχρέωση να τις τηρήσουμε. Εάν δεν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες, τότε η εμπιστοσύνη του κόσμου μειώνεται. Αυτό αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι μπορέσαμε να εγκρίνουμε, μάλλον εγκρίθηκε δηλαδή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ήδη πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εάν ήμασταν υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με προσωρινούς προϋπολογισμούς, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά μας. Όμως όπως είπαν ήδη άλλοι, η κρίση αυτή πληρωμών, γύρω από τις πληρωμές δηλαδή, δεν είναι τίποτα το νέο. Έχει αρχίσει από το 2011. Δυστυχώς, 80% των καθυστερήσεων στις πληρωμές πλήττει την πολιτική συνοχής. Μα αυτή η πολιτική συνοχής όμως στοχεύει στη μείωση των αποστάσεων μεταξύ των χωρών μελών. Η πολιτική συνοχής είναι από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα έχει απτά αποτελέσματα, αποτελέσματα τα οποία είναι και ορατά όταν δει κανεί και τις αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια. Εκεί βλέπουμε πραγματικά τις αλλαγές που επέφερε η πολιτική συνοχής. Αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές θίγει κυρίως τους δικαιούχους έργων επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων. Η πολωνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα, έδωσε προκαταβολές στη βάση των ε, δεσμεύσεων που είχαν αναλυθεί για, το, τη 2007 έως 2014 περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ και στην παρούσα περίοδο 2014 έως 2020 θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική Τώρα όμως έχουμε δύο φορές λιγότερες, λιγότερες προκαταβολές σε αυτή την περίοδο. Η πολωνική κυβέρνηση θα χρειαστεί λοιπόν να πληρώσει από το δικό της τον εθνικό προϋπολογισμό τους δικαιούχους των κοινοτικών επιδοτήσεων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας και στη σχέση μεταξύ ε, κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εντύπωση που έχουμε όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύει τις πληρωμές, τις μπλοκάρει χωρίς επαρκή αιτιολογία. Και όμως λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις συνεισφορές των χωρών μελών. Και οι χώρες μέλη έχουν όλο και περισσότερες δυσκολίες να πληρώσουν αυτές τις συνεισφορές. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει διορθώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς κάθε φορά που έγιναν αλλαγές τις υποστηρίξαμε διότι αντιλαμβανόμαστε υπάρχει ανάγκη να ε, εκπληρούνται οι υποχρώσεις ιδίως μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους καθαρούς εισφορείς ήταν ανάγκη, η ανάγκη να πληρώσουν ακόμη περισσότερο ως συνεισφορές για να ξεπεραστούν αυτές οι διαφορές μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν ωστόσο η συνεισφορά της Μεγάλης Βρετανίας. Εν ώψη του μεγέθους της συνεισφοράς αυτής, πολλές ε, κυβερνήσεις χρειάστηκε ε, να ε, προσφύγουν σε δόσεις, σε καταβολή σε δόσεις της συνεισφοράς τους. Όπως είπε προηγουμένως η Ευρωπαία Επίτροπος, το κλείσιμο των λογαριασμών της προηγούμενης περίοδου, θα, από αυτό μάλλον θα προκύψουν και άλλες υποχρεώσεις πληρωμών. Και ταυτόχρονα θα έχουμε και αύξηση των πιστώσεων υποχρεώσεων λόγω των νέων έργων που πάνε τώρα να εγκριθούν για την επόμενη περίοδο. Έχουμε και την ιστορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, βεβαίως και την κατάσταση στην Ελλάδα που θα χρειαστεί περισσότερη την προσοχή μας. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι απολύτως απρόβλεπτη. Δεν ξέρουμε πώς θα χρειαστεί να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως σε μια ένταση του ρωσικού εμπάργου. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι η κατάσταση θα αντιμετωπίζεται καλύτερα στο μέλλον και ότι θα τεθεί υπό έλεγχο παρόλες τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που εντείνει την ανησυχία μας. Άλλη ε, κατάσταση που εντείνει τις ανησυχίες μας είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι πρέπει κανείς να ξεπλώνει τα χρέη του για μας είναι προφανές. Θέλουμε όλες οι χώρες μέλη να σκέφτονται βεβαίως το ίδιο. Η κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Joint Statement που έχει προσαρτηθεί στον ε, Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό μας δίνει κάποιες ελπίδες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι χώρες μέλη θα καταβάλουν, θα εκπληρώσουν τις υποχρώσεις τους. Και τώρα, για να δούμε πώς ε, πραγματώνεται, υλοποιείται αυτή η πραγματικότητα, θα ακούσουμε τον κύριο Ζαν Νοελ Γκότιε, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρώπη και Διεθνή Στρατηγική, που είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο της περιοχής του Λίγυρα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρτουή για την πρόσκλησή του και την ευκαιρία που μου δίνει να σας δείξω επιτόπια τι σημαίνει καθυστέρηση πληρωμών. Θα ήθελα να πω ότι είμαι υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχήν. Δεν θα μιλήσω εξ ονόματος μιας περιφέρειας, αλλά εξ ονόματος ε, της Ευρώπης, που εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη περιοχή, διότι εμείς, ε, όπως καταλαβαίνετε, Είμαστε ο τελευταίος τροχός της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εμείς θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την στρατηγική για να κατανοήσουν και οι πολίτες τι σημαίνει. Πρόκειται μεγάλη, για μεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά. Η περιφέρεια του Λίγυρα, όπως ξέρετε, για την περίοδο 14-20 έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ως περιφέρεια και θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα της Ευρώπης. Και αυτό χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία υπάρχουν, πληθώρα αυτών υπάρχει, αλλά υπάρχουν δυσκολίες και αυτό αφορά την κακή εικόνα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωση στον τομέα. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Αρτουίν να μπορέσω να σας μιλήσω για αυτά τα δεδομένα για να σας πω ε, πώς έχει το ζήτημα σε εθνικό επίπεδο. Ως προς την περίοδο 7-13 θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς ε, έγιναν τα πράγματα. Όπως ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση η νομαρχία ήταν υπεύθυνη για την διαχείριση των κονδυλίων και θα έπρεπε να γνωστοποιήσει τις προβλέψεις ως προς τις πιστώσεις πληρωμών. Το 2012 ήδη γνωρίσαμε καθυστερήσεις ως προς τις επιστροφές του ΕΤΠΑ Ε, πρόκειτο για ε, διαγωνισμούς που έγιναν στις, ε, στα τέλη του 12 για την περίοδο 12-13 και είχαμε καθυστέρηση 144 ημερών για την καταβολή των ποσών. Άρα δεν τηρήθηκε ο κανονισμός του 2006, το άρθρο 87 που αναφέρει ότι τα κονδύλια αυτά πρέπει να καταβληθούν μέσα σε δύο μήνες. Παράλληλα, είχαμε διακοπή πληρωμών στην αρχή του 2012 μετά από ελέγχους που αφορούσαν ολόκληρη τη Γαλλία. Όπως καταλαβαίνετε, η καθυστέρηση αυτή και η διακοπή πληρωμών, η πάυση πληρωμών, δημιούργησε μεγάλα οικονομικά προβλήματα διότι οι δημόσιες αρχές δεν μπορούν να προωθήσουν ε, αυτό το ευεργέτημα, αυτές τις πληρωμές ε, στο, στους ε, δικαιούχους και επίσης αυτή η κατάσταση δεν είναι ευεργετική ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια των παρεμβάσεων της Ευρώπης υπέρ των πολιτών. Εκείνη την περίοδο δεν ήμασταν παρά ενδιάμεση για τη διαχείριση των ε, λογαριασμών αυτών, μιλώ για την περιοχή του Λίγυρα, έπρεπε όμως να προωθήσουμε συγκεκριμένα κονδύλια για να μην υπάρξουν δυσκολίες ε, στην ανάληψη έργων. Μιλήσαμε για την περίοδο 7-13. Θα ήθελα να επιμείνω έτσι ώστε η περίοδος 14-20 να μην γνωρίζει τέτοιες δυσκολίες. Και αυτό από, αφορά όλες τις περιφέρειες της Γαλλίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μία προπληρωμή εμείς και να έχουμε καθυστέρηση καταβολής των πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών. Ο κύριος Αρθή μίλησε για την Ευρώπη η οποία λεπτολογία. Αυτό το ζούμε καθημερινά. Και αυτό αφορά τους επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε εθνικό επίπεδο για σχέδια τα οποία δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, που απλώς συγχρηματοδοτούνται από την Ευρώπη και αυτό ειδικά την περίοδο 7-13. Γι' αυτό θα ήθελα να τηρηθούν οι προθεσμίες ε, καταβολής πληρωμών. και η κατάρτιση των φακέλων είναι μία πολυσχηδής ε, διαδικασία και αυτό αφορά και τις διαχειριστικές αρχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ την ανάγκη ελέγχων για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά θα ήθελα να σας τονίσω ότι υπάρχει ένα χρονικό χάσμα μεταξύ των πληρωμών και των άμεσων αναγκών των δικαιούχων. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, σύστημα προπληρωμών αρχικών δηλαδή καταβολών σε τοπικό επίπεδο, αλλά το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Επιτροπής δεν το επιτρέπει με στα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης και της ε, ανάληψης υποχρεώσεων. Χωρίς λοιπόν αυτή την ε, συνέχεια στους δικαιούχους, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν ε, κίνητρα έτσι ώστε να προωθηθούν συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα. Διότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι και ένας παράγοντας προώθησης προγραμμάτων. Εάν οι μικροδικαιούχοι προβάλλουν προγράμματα μικρής ενδέλειας και κλίμακας, εάν δεν έχουν αυτή την χρηματοδότηση δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, διότι οι μικροί αυτοί παράγοντες θα μπορέσουν να προωθήσουν την πραγματική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας δώσω δύο απτά παραδείγματα που χρειάστηκε να διαχειριστούμε σε επίπεδο ε, τεχνικής, τε, τοπικής αυτοδιοίκησης το ένα ε, συγκεκριμένο πρόγραμμα που, όπου συμμετείχαν ε, οι βιομηχανίες και οι ακαδημαϊκοί κύκλοι, το μικροκομπούς, το οποίο προωθήθηκε σε τοπικό επίπεδο και αφορούσε 41 εκατομμύρια η τελευταία πληρωμή μέσα στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης έγινε το 2014, δηλαδή 7 χρόνια μετά από την υποβολή του φακέλου. Επίσης, ως προς τη γραμμή Νόνσα Τομπριόν, σιδηροδρομική σύνδεση, το Μάρτιο του 2011 υποβλήθηκε το σχέδιο και τώρα έχει καταβληθεί το 60% ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση ισχύει εδώ και ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο πλαίσιο συνδιαχείρισης και πολλές φορές η διαχείριση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν οδηγεί σε ένα γραφειοκρατικό και διοικητικό φόρτο. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι επειδή μιλήσαμε για ελλείμματα και ελλείψεις θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι τοπικές αρχές έχουν να επομιστούν ένα μεγάλο οικονομικό βάρος και το 75% του άχθους αυτού το επομίζονται οι τοπικές αρχές. Κατανοούμε τους ελέγχους, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι παύσεις πληρωμών και οι καθυστερήσεις δημιουργούν στενοπούς, κάτι το οποίο επιβαρύνει τις τοπικές αρχές. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρήσουν τους μακροοικονομικούς όρους που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για τη διαχείριση του, των ελλημάτων. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια χρυσή τομή, αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας βοηθήσετε και οι πολίτες δεν μπορούν να διακρίνουν και να επιμερίσουν τις ευθύνες. Η Ευρώπη αποτελεί ένα σύνολο για τους πολίτες και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επιλύσουμε από κοινού αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν την καταβολή των επιδοτήσεων. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του κυρίου Αρτουή. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα και η περιοχή του Λίγυρα θα συνδράμει στις συγκεκριμένες εργασίες με, τις επιτόπιες, ε, με την επιτόπια πείρα μας και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε επίπεδο περιφερειών έτσι ώστε να συμφιλιώσουμε την Ευρώπη με τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνδρομή σας και μιλήσαμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σάντος Γιόρνα, ο οποίος είναι δήμαρχος της Αρόγιο Ντελαλούθ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, Ειλικρινά ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την ε, πρόσκληση που μου απέστειλε. Για να σας προσφέρω την άποψη ενός δήμαρχου, ενός ε, δήμου της Ισπανίας, του Αρόγιο Ντελαλού, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς τα χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια σήμερα. Θέλω επίσης να σας προσφέρω και τις εντυπώσεις που έχω για ενδεχόμενε αλλαγές που θα σύστηνα να γίνουν για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση και χρήση των ευρωπαϊκών αυτών κονδυλίων. Εννοείται ότι σας συγχαίρω για την ιδέα σας, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω απ' όλα, να κάνει συζήτηση για αυτό το θέμα το οποίο επηρεάζει τους πολίτες, τους δήμους μας. Είναι καλό που συμμετέχουν λοιπόν και οι Δήμοι στη συζήτηση αυτή, γιατί οι Δήμοι είναι αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη. Θέλω λοιπόν να σας παρουσιάσω το μέρος από το οποίο προέρχομαι. Το χωριό, το οποίο είμαι εγώ δήμαρχος, που ονομάζεται Αρόγιο Ντελαλούθ, είναι ένα μικρό χωριό με 1.400 κάτοικους που βρίσκεται στην Εξτρεμαδούρα, μια ισπανική περιφέρεια η μοναδική σύγκληση σήμερα στόχου 1 και δεν πρόκειται, για τους, δεν πρόκειται για το πιο μικρό δήμο, θα έλεγα από τους πιο μεγάλους της Εξτρεμαδούρα. Μιλάμε λοιπόν για το αρρώγιο Ντελαλούθ, μιλάμε για την πραγματικότητα που ισχύει σε πάρα πολλού Δήμου, ολόκληρη την Ισπανία, αλλά σίγουρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Πέρυσι λοιπόν είχαμε ένα ρεκόρ το 2014 και δεν ξέρω αν σα φαίνεται σημαντικό ή όχι, εγώ το βρίσκω σημαντικό. Γεννήθηκαν 53 παιδιά. Πριν από 13 χρόνια δεν είχαμε τόσα πολλά παιδιά να γεννιούνται στο χωριό μας, κάτι το οποίο μας δίνει ελπίδα για το μέλλον. Και το πρώτο δώρο που παίρνουν τα μωρά αυτά είναι ε, μια κάρτα ε, μέλους στην ε, τοπική μας βιβλιοθήκη. Στο Αρόγιο Ντε Λαλούθ είχαμε και εμείς κρίση που μας χτύπησε πολύ από το 2007 μέχρι το 2014 επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των ανέργων. Ήμασταν γεωργικός δήμος, κτηνοτροφικός πριν από λίγο, ενώ τώρα αφιερώμαστε ασχολούμαστε με, την, με τις οικοδομές, τον οικοδομικό τομέα. Η ανεργία μας έπληξε πάρα πολύ και η καταπολέμησή της είναι ο πρώτος μας στόχος. Κάτι το οποίο ισχύει βέβαια σε πολλούς δήμους της Ευρώπης. Εμείς θέλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς πολίτες, να ζούμε αξιοπρεπώς, με ισότητα ευκαιριών και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξηγώ τι εννοώ. Ήταν πολύ σημαντικό για το Δήμο μας να έχει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με τις προσπάθειες του Δήμου μας αλλάξαμε το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής και βοηθήσαμε νέους και μεγαλύτερους. Με κατάρτιση 500 ακολουθούν επιμόρφωση. Με τη βοήθεια επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κονδύλια από το Δήμο στοιχηματίζουμε υπέρ της οικολογικής και πράσινης γεωργίας. Φτιάξαμε την πρώτη τράπεζα γεών. Προκειμένου οι καταλελειμμένες γεές να δοθούν δωρεάν σε νέους για να τις δουλέψουν. Με τη βοήθεια του Δήμου αρχίσαμε να λειτουργούμε και τον πρώτο συνεταιρισμό νέων που πουλούν απευθεία στον καταναλωτή τα φρούτα τους και τα προϊόντα του με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κονδύλια από το Δήμο μα. Τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε και κοινωνικές υποδομές που δεν είχαμε πριν. Νηπιακό σταθμό, ε, για άτομα που δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους σε ένα κέντρο για να περνάνε τη μέρα Δίνουμε κοινωνική προσοχή δηλαδή κατά προτεραιότητα σε αυτού που έχουν ανάγκη και δημιουργούμε συγχρόνω και θέσεις απασχόληση. Με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κονδύλια από το Δήμο μα επίση. ο πολιτισμό και ο αθλητισμός έγιναν δικαίωμα και όχι πολυτέλεια για το Δήμο μα Πάνω από χίλιοι είναι γραμμένοι στο τοπικό κέντρο και κάθε Κυριακή έχουμε εκδηλώσεις, κινηματογράφο με ταινίε. Ξαναφτιάξαμε τον κινηματογράφο και σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι οι νέοι μπορούν να έχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις και να αθλούνται σε καθημερινή βάση. Μπορεί να ακούγεται ψέματα πως ένας δήμος 1400 ε, ε, πολιτών, κατοίκων να έχουν μια ομάδα αθλητική η οποία να βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα αν τη συγκρίνουμε με άλλες στη χώρα, στην δεύτερη κατηγορία. Ο Δήμος, επίσης, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε τη συμμετοχή των πολιτών βασικό στοιχείο για την τροποποίηση του Δήμου μας. Έχουμε ένα κέντρο επίσης για τους ηλικιωμένους όπου αποφασίζουν οι πολίτες. Συμμετέχουν και επιχειρήσεις. 100 επιχειρήσεις περισσότερες έχουμε σήμερα από ό,τι την περίοδο που άρχισε η κρίση. Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε με 11.000 ευρώ να βοηθήσουμε στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων αυτών και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Κατάρτιση επίσης για τους άνεργους, όπως σας είπα, νέες κοινωνικές υποδομές όπου έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Σήμερα πρέπει να δουλέψουμε και υπέρ της ένταξης όλων των πολιτών. Να μην υπάρχει καμία οικογένεια στο Δήμο μας που να μην έχει είτε ηλεκτρικό, είτε τρόφιμα, είτε νερό, είτε σπουδές. Κανείς να μην χάνει και κανείς να μην χαθεί στο δρόμο. Ο δρόμος σίγουρα ήταν δύσκολος τα τελευταία 12 χρόνια. Εμείς βελτιώσαμε τις κοινωνικές υπηρεσίες και να ξέρετε ότι ο Δήμος μας δεν έχει κανένα δάνειο και κανένα χρέος. Αυτό το οποίο κάνουμε με τις προσπάθειές μας που είμαστε όπως σας είπα ένα μικρό χωριό από μία περιφέρεια στόχου 1 της σύγκλησης σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να πετύσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους υπόλοιπους να κάνουν τις ίδιες προσπάθειες όπως κάναμε και εμείς. Στον αγώνα αυτό όμως, τον οποίο δεν σταματάμε, υπέρ των ε, δημοτών μας, πρέπει να ξέρετε ότι συναντήσαμε και εμπόδια, τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε και θα σας τα εξηγήσω. Σήμερα λοιπόν καταγγέλουμε πώς είναι δυνατόν στην κατάρτιση των ανέργων τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάνουν με τόσο μεγάλη καθυστέρηση και έτσι να μην μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τους μαθητές ούτε τους δασκάλους. Την τελευταία φορά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο που μας πέρασε του 2014 με χρήματα από την κυβέρνηση της ε, Εξτραμαδούρα και από την εγγύηση το, για την νεολαία έπρεπε να πληρώσουμε τους νέους. Σήμερα λοιπόν κατακέλω πώς είναι δυνατόν η εφαρμογή της πράσιμης ανάπτυξης με ευρωπαϊκά κονδύλια τελικά από την Ευρώπη να πάρουμε τα χρήματα ένα χρόνο αφού είχαμε ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να χρεωθεί ο Δήμος για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο. Σήμερα καταγγέλω εδώ και σας ρωτώ πώς είναι δυνατόν ένα οικονομικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόθεση της υγείας, την πρόληψη δηλαδή, για να ενισχυθούν οι οικογένειες, τα παιδιά στο χωριό μου όπου σε συνεργασία με την Νορβηγία, τη Δανία κλπ. να μπορούμε να έχουμε 60% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τελευταία πληρωμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει γίνει μέχρι τον Νοέμβριο του 2014. 1,5 χρόνο δηλαδή αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα το οποίο καθημερινά εφαρμόζεται σε ένα σωρό δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγγέλλω λοιπόν εδώ και σας ρωτάω πώς είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα για το εμπορικό επιμελητήριο που χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλει το επιχειρησιακό επίπεδο του χωριού μου σε ένα ανώτερο επίπεδο να καταλήξει να πρέπει ο Δήμος να προκαταλάβει τα χρήματα γιατί δεν έχουν γίνει πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έπρεπε και να καλύψουμε έτσι εμείς τα χρήματα που έπρεπε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πραγματικότητα η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά σε ένα σωρό δήμου τη χώρα μου. Καταγγέλλω εδώ σήμερα λοιπόν και σα ρωτώ πώ είναι δυνατόν η δίκηση που διαχειρίζεται τα περιφερειακά κονδύλια προ την αυτόνομη περιοχή τη Εξτρεμαδούρα να καθυστερούν τόσο πολύ για τι πληρωμέ που γίνονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία που καταλαβαίνετε τι σοβαρά προβλήματα δημιουργεί στα δικά μας ταμεία και στα προγράμματα τα οποία εφαρμόζουμε με τα χρήματα αυτά. Κάτι το οποίο ισχύει και στο δικό μου Δήμο αλλά και σε ένα σωρό άλλους. Εν κατακλείδη. Το Ρόγιο Ντελαλουθ, όπω και τόσοι άλλοι δήμοι στην Εξτρεμαδούρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για να δώσουμε όθηση στου πολίτε μα για να του δώσουμε περισσότερε ευκαιρίε στην κατάρτιση και στην απασχόληση από ό,τι κατά το παρελθόν. Με το στόχο αυτό τα Ευρωπαϊκά Ταμεία με χρηματοδότηση αϊφόρου ανάπτυξης είναι κάτι αναγκαίο σε μια περιφέρεια προτεραιότητας όσον αφορά τη σύγκληση, την εξτρεμαδούρα. Τα χρήματα αυτά όμως, τα κονδύλια αυτά δεν φτάνουν στους τελικούς δικαιούχους κάτω από τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες και οι λόγοι είναι πολύ και διάφοροι. Πρώτον, οι εθνικές αρχές πολλές φορές καθυστερούν να πληρώσουν τις περιφερειακές αρχές και έτσι δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητα και λογιστικό πρόβλημα. Δεύτερον, οι περιφερειακέ αρχές πολλέ φορέ στέλνουν στους τελικού δικαιούχους, είτε είναι αυτοί οι δήμοι, είτε κοινότητε, είτε επιχειρήσει, είτε οργανώσει, πολύ αργά τα χρήματα, με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, το οποίο οδηγεί σε προβλήματα ρευστότητα και λογιστικά. Μεγάλα προβλήματα έχουν οι Δήμοι όταν ξεκινούν προγράμματα ευρωπαϊκά, αλλά τα κονδύλια δεν φτάνουν όταν θα έπρεπε να φτάσουν έτσι όπως έχει συμφωνηθεί. Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερούν τα χρήματα και στον τελικό δικαιούχο. Πολλές φορές υλικά δεν είναι δυνατόν οι Δήμοι να καλύψουν αυτή την έλλειψη κονδυλίων. Το γεγονός ότι πρέπει εμείς να δίνουμε προκαταβολές, μερικές φορές να χρηματοδοτούμε πλήρως προγράμματα, εμείς οι Δήμοι, επειδή δεν έχουν έρθει τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σαν αποτέλεσμα πολλά, πολύ, πάρα πολλοί δήμοι τελικά να απορρίπτουν προγράμματα συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορούν να το επιτρέψουν στον εαυτό τους να αναλάβουν αυτή το κόστος. Όταν αποφασίζουν κάποιοι να επενδύσουν στους δήμους, πάρα πολλές φορές διαπιστώνουν ότι τα κριτήρια δεν είναι όπως είχαν καταλάβει στην αρχή, ότι μερικές φορές τα κριτήρια είναι περισσότερο πολιτικά και τελικά τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά δεν φτάνουν στους Δήμους έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει διαφάνεια, συνεπώς, για τον τρόπο με τον οποίο επενδύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή πού πάνε τελικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η αξιολόγηση της χρηματοδότησης να μην γίνεται όπως πρέπει και να μην ξέρουμε ποια είναι ακριβώ η κατάσταση και τελειώνω. Εξαιτία όλη αυτή τη προβληματική που πλήττει Δήμου σαν το δικό μου, ε, Δήμου τη χώρα μου, Δήμου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να τελειώσω με κάποιε συστάσει, όσο μου επιτρέπεται, για νέα λειτουργικά προγράμματα. Είναι αναγκαίο απαραίτητο να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση που να καθορίζει τις προθεσμίες και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στους δικαιούχους τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πώς θα χρησιμοποιούνται επίσης από τους δικαιούχους, όπως είναι οι Δήμοι, να απαιτούνται συγκεκριμένες προθεσμίες όσον αφορά τις πληρωμές. Δεύτερον, να μην υπάρχουν αυθαίρετα συστήματα. Οι Δήμοι να μην πρέπει να προκαταβάλουν τα χρήματα, είτε το μεγαλύτερο μέρος, είτε το σύνολο των επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν να υπάρχουν προκαταβολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα. Τρίτον, πρέπει να μειωθούν οι προθεσμίες για την πληρωμή των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τους Δήμους. Άπαξ και οι Δήμοι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τότε πρέπει να πληρώνονται. Δεν πρέπει να υπάρχουν καθυστέρησεις, να μην αργεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, θα πρέπει να υπάρχει ελεγκτικό σύστημα ώστε οι εθνικές και περιφερειακές αρχές όταν επενδύουν με ευρωπαϊκά κονδύλια στους διάφορους δήμους να υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι και προτεραιότητες για τα λειτουργικά προγράμματα. Πέμπτον, πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο και να έχουμε μηχανισμούς διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής των πολιτών και στο σχεδιασμό των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και στην κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων δήμων. Να συγκρίνουμε ποια είναι η αναγκαιότητα κάθε φορά και να συγκρίνουμε και με άλλες περιοχές. Επίσης πρέπει να παρακολουθούμε πώς γίνονται οι πληρωμές και των ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και τη χρηματοδότηση από το εθνικό, το περιφερειακό ή το, κοινοτικό, το δημοτικό επίπεδο. Να γίνεται περιοδική αξιολόγηση επίσης των πληρωμών που έχουν γίνει σε κάθε Δήμο για να διαπιστώσουμε ποια ακριβώ είναι η καθυστέρηση για κάθε πρόγραμμα και ποιο είναι το επίπεδο εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στο πρόγραμμα. Να αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του και ο καθένας να <clears throat> ξέρουμε πόσο φταίει, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται. Αν υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία φτάνουν στο Δήμο μου μέσω ε, τοπικών ε, οργανώσεων, μέσω του Leader ή οτιδήποτε και περνάει χρόνος, ένας μήνας, ενάμιση μήνας, καταλαβαίνετε ότι αυτό καθυστερεί άλλα προγράμματα αν δεν έχουμε πάρει τα χρήματα και συσσωρεύεται η καθυστέρηση τελικά στις πληρωμές. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να γυρνάμε και να κοιτάμε από την άλλη μεριά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Όταν ένας Δήμος δεν μπορεί να πληρώσει τους ε, εργαζόμενούς του επειδή δεν έχουν έρθει ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ε, το πρόγραμμα το οποίο κανονικά πρέπει να πληρωθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια, καταλαβαίνετε ότι καθυστερεί πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιο σφάλμα εδώ. Αν δεν μπορεί να συμμετέχει ένα Δήμο σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, επειδή πρέπει ο ίδιο να πληρώσει τη χρηματοδότηση που κανονικά πρέπει να έρθει από την Ευρώπη. Σήμερα στο Ρόγιο Ντε Λαρούθ, στου Δήμου τη Εξτραμαδούρα, τη Ισπανία και τη Ευρώπη, χρειάζεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να ενισχυθεί η του κόσμου και να αποκατασταθεί αυτή αυτή η χρηματοδότηση δεν μπορεί να καθυστερεί ή να μην φτάνει ποτέ. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, να υιοθετηθούν μέτρα, να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν τα εκατομμύρια των πολιτών που ζουν σε μικρούς και μεσαίους δίπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και σας ζητάω παρακαλώ να έχετε το θάρρος που όπως έχουν και οι δήμαρχοι την ε, χώρα μου και στην Ευρώπη ολόκληρη, ώστε να ανακτήσουν αξιοπρέπειά τους οι πολίτες και του δικού μου Δήμου, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χώνα. Δύο διευκρινήσεις. Μέχρι το τέλος της συνεδριασής μας θα εξακολουθήσουμε να έχουμε διερμηνία προς τα Μαλτέζικα, αλλά η κυρία Επίτροπος θα πρέπει να φύγει στις 12.45 και δεν είναι εύκολος ο ρόλος σας, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό γιατί οι κυβερνήσει αναλαμβάνουν υποχρέωση μετά δεν πληρώνουν. Και η Κομισιόν προσπαθεί να εξασφαλίσει κάποια συνεκτικότητα μεταξύ πληρωμών και υποχρεώσεων. Οι μαρτυρίες που ακούσατε δείχνουν την ανάγκη να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια από την πλευρά των κυβερνήσεων που δεν μπορούν να παραμείνουν στην αμφισημία. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε, πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο λεπτά μάξιμουμ παρακαλώ, δύο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα βρήκα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν και από την ε, πλευρά της Επιτροπής Ελέγχου του που προεδρεύω είναι το καθημερινό μας ψωμί και βούτυρο. Είμαι από το θέλω να σα αναφέρω ορισμένα προβλήματα που έχουμε δει ήδη από το 2013. μα. ενοχλεί πολύ ότι δεν λειτουργεί καλά το σύστημα ελέγχου στα κράτη-μέλη και θέλω να εστιάσω την προσοχή σα στο σημείο αυτό και να σα παρακαλέσω να σκεφτείτε και να εργαστείτε λίγο περισσότερο για το θέμα αυτό γιατί έχει σημαντικέ επιπτώσεις στον τομέα του προπολογισμού. Στη Γεωργία, στα μέτρα για την Ήπεθρο, έχουμε θέση σε κίνδυνο πάνω από 2 εκατομμύρια για τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλιστούν αυτά τα κονδύλια στον τομέα της, των εγγύσεων έχουμε περάσει τα 56 εκατομμύρια στην ε, Γαλλία, 18 στη Γερμανία, 17 στην Ελλάδα, 200 στη Γαλλία. Αυτά είναι θέματα άμεσων πληρωμών. 600 εκατομμύρια έχουν τεθεί σε κίνδυνο και αυτό σε 19 κράτη-μέλη της Ευρώπης. Δεν έχουν εξασφαλιστεί οι πληρωμές αυτές. Έχουμε συνολικά και στον τομέα των διαφθορτικών τομέων έχουμε 440 εκατομμύρια τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο. Παίρνουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη που δεν είναι <clears throat> απόλυτα ακριβή. Και βλέπει η Κομισιόν ότι υπάρχει ένα επίπεδο σφαλμάτων που για τα κάτι μελη είναι 0,6% ενώ για την Κομισιόν είναι 5,6%. Όλα αυτά είναι σημαντικέ τροποποιήσει που δεν μπορούμε να τι παραγνωρίσουμε. Γι' αυτό σα παρακαλώ να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια για τον ελεγκτικό σύστημα και επίση για τα μέσα χρηματοοικονομικής μηχανικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πληρώσει σημαντικά χρήματα σε τράπεζε στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την ε, Λιθουανία, την ε, Ιταλία και την Ελλάδα που δεν έφτασαν ποτέ τον τελικό τους δικαιούχο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω, επειδή είναι σαφές και από την έκθεσή μου, ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και νομίζω ότι και αυτά που ελέγχθησαν από τις προελίσσαντες είναι σαφή. Γι' αυτό κάντε κάτι <clears throat> για να υπάρξει πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου στα κράτη-μέλη, το οποίο έχει φανεί ότι είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Ήδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Χρειάζεται έλεγχος, αλλά δεν πρέπει να πολυπλοκοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα. Ο κύριος Πράγμαν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν κινδυνεύει μόνο η αξιοπιστία όταν δεν πληρώνει κανείς τους λογαριασμούς του. Τίθεται και το ερώτημα εάν με το πλήθος των διαφόρων έργων που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές είτε από το ε, Γεωργικό Ταμείο είτε από το Περιφερειακό Ταμείο και ούτω καθεξής όπου εν τέλει μιλούμε και για επιδοτήσεις λιγότερες των 100.000 ευρώ όλα αυτά λοιπόν δεν, δεν ε, πληρώνονται, πολλοί από τους λογαριασμούς αυτούς που δεν, που δεν πληρώνονται και το ερώτημα είναι εάν ίσως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαμορφώνει τα προγράμματά της έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερα και να ανταποκρίνονται τις ανάγκες που συζητήσαμε και σήμερα το πρωί σε Ολομέλεια. Να είναι δηλαδή μια ορατή συμβολή ως ανθρωπιστική ενίσχυση ή για τη βελτίωση των υποδομών. Κάνω λοιπόν το εξής σύντομο σχόλιο. Ακούστηκε πριν ότι οι πόροι αυτοί πρέπει να προσφέρουν αξία. Εάν πρέπει να προβλέπεται η χρηματοδότησή τους εθνικούς προϋπολισμούς για να λαμβάνουν και τη χρηματοδότηση, τότε πρέπει να ανοίγουν και την δυνατότητα χρηματοδότησης από τα εθνικά κοινοβούλια. Και τέλος η διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Καλύτερα να στοχεύει συγκεντρώνονται οι πόροι και να στοχεύονται εκεί όπου αποδίδουν. Αυτό νομίζω θα αυξήσει και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά, σημαντικά μάλιστα, και ταυτόχρονα θα μειώσουν την επίπτωση της μη, πληρωμή, πληρωμής λογαριασμών σε θέματα αξιοπιστίας. Ο κύριος Ντεμονγκολφιέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, γιατί θέσατε αυτό το θέμα επιτάπητος. Γίνεται λόγος για 23 δις ευρώ και τις δυσκολίες που έχουν οι τοπικές αρχές να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την πληρωμή με βάση τις καθυστερήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν ως προς το διακύβευμα αυτό και τις διαφορές. Ε, υπάρχουν ε, διαφορές ε, σε σχέση με τα μη καταβληθέντα ποσά. Πώς έχουμε διευθετήσει αυτό το θέμα των ενδεχόμενων διαφορών ως προς την καθυστερημένη καταβολή πληρωμών. Έχουμε πληροφορίες για τα μεγάλα προγράμματα, αλλά μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις καθυστερήσεις πληρωμών. Ο κύριος Σίγφριντ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε διότι θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Αλτουή διότι μας επεξήγησε πώς έχουν τα γεγονότα και μας επεξήγησε επακριβώς την κατάσταση διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο. Φτάσαμε στο τέλος σε μια συμφωνία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Βεβαίως υπάρχουν ε, απλήρωτοι λογαριασμοί ακόμα και σήμερα, κάτι το οποίο δείχνει ότι θα πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά. Πέρσι καταφέραμε, όπως είπατε σωστά κυρία Πίτροπε, να σταθεροποιήσουμε το θέμα, αλλά δεν φτάσαμε σε μια βιώσιμη λύση και η δημοσιονομική κρίση που αποφύγαμε το 2014 ίσως ε, πραγματοθεί φέτος ή του χρόνου με βάση τα παραδείγματα που είδαμε διότι δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε το 14 και στις αρχές του 2015. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς ε, μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο να βρούμε μία μακροχρόνια λύση στο θέμα των πληρωμών και αυτό μπορεί να αφορά ένα σύστημα ίδιων πόρων που να είναι απλό, αδιαφιλονίκητο και ε, διαφανές. Δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύετε ότι μία μακροχρόνια λύση μπορεί να εξευρεθεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας ε, θητείας και ποια είναι η θέση της Επιτροπής για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων για να επιλύσουμε αυτό το θέμα των ανεπαρκιών στις πληρωμές, αν λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές σχέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων με τις κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφέρω τη γνώμη μου στο Κοινοβούλιο που εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη. Να σας μιλήσω για τη θέση της Ισπανίας, η οποία βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση Έγιναν πολλές συζητήσεις και σήμερα το πρωί για την ενδεχόμενη συμβατότητα των πολιτικών λιτότητας με μια πολιτική απασχόλησης και ανάπτυξης. Θα ήθελα να τονίσω την προσπάθεια που έκανε η Ισπανία για να καταβάλει τα χρέη της, για να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της και να συνδυάσει αυτό αυτή τη δέσμευση με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες αλλάζουν την οικονομική κατάσταση. Η Ισπανία γνώρισε οικονομική ύφεση, αλλά βρίσκεται επικεφαλής της Ευρώπης σε οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας χάρη σε αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μέσα στα πλαίσια και της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι έχουμε ανταποκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει παράλληλα με την ε, δημοσιονομική αυτή ε, ολοκλήρωση να δώσουμε ε, νέα κίνητρα για μια πολιτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, θεώρηση που μας έδωσε ο Δήμαρχος από την Ισπανία, έτσι ώστε τα διαρθρωτικά ταμεία να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στη χώρα μας, στην Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, και ο Πρόεδρος. Λόγω της πίεσης χρόνου της κυρίας Επιτρόπου, η οποία θα πρέπει να φύγει σε 7 λεπτά, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε στην πρώτη σειρά ερωτήσεων που σας έχουν τεθεί. Ευχαριστώ και εκφράζω τη λύπη μου που είμαι υποχρεωμένη να σε εγκαταλείψω εντός ολίγου. Έχω άλλη ανηλυμένη υποχρέωση συνάντηση με μια ομάδα γυναικών και νομίζω ότι θα είναι έλλειψη σεβασμού εάν δεν εμφανιστώ να τη συναντήσω. Σε παρένθεση τώρα, ένα από τα καθήκοντά μου ως αντιπροέδρου για αρμοδίας για ανθρωπίνους πόρους είναι και να φροντίσω να συνεχίσουμε τον στόχο, την επιδίωξη του στόχου το να βάλουμε 40% γυναίκες στην Κομισιόν για να πετύχουμε μεγάλη αποδοτικότητα και απόδοση. Μικρή υποσημείωση. Με ενδιαφέρον παρακολούθησα στα σχόλια του Ισπανού Δημάρχου πόσο σημαντικού, σημαντική για αυτό είναι να περιλαμβάνονται όλοι οι συμπερίληψη δηλαδή και έτσι έχουν και ποδοσφαιρικές ομάδες ανδρών και γυναικών. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως, το πρώτο που ακούστηκε σήμερα ήταν και το πιο σημαντικό νομίζω κρισιμότητα δηλαδή της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Σχέση εμπιστοσύνης δηλαδή με τους πολίτες. Η αξία της Ευρώπης, η αξιοπιστία της Ευρώπης και βεβαίως το θέμα της αποπληρωμής των λογαριασμών είναι τμήμα αυτής της προσπάθειας αποκατάστασης εμπιστοσύνης και όχι μόνο για τα μεμονωμένα επιδοτούμενα έργα, για το γενικότερο καλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουμε αυτό το θέμα του να κατεβάσουμε δηλαδή αυτή την μη πληρωμή των λογαριασμών σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο όχι αργότερα το 2016, το παίρνουμε λοιπόν αυτό πολύ στα σοβαρά. Τώρα, έχω να σας κάνω τέσσερα σχόλια εις απάντηση των δικών σας. Πρώτο, καθυστερήσεις. Άκουσα δραματικές περιγραφές καθυστερήσεων που δώσατε και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, κάποιος θίγεται. Μπορεί να είναι μια επιχείρηση, μπορεί να είναι ότι πρέπει να πληρώσουν τόκους, μπορεί να είναι ένα φορολογούμενος. Αλλά οι καθυστερήσει, δυστυχώ, τυχαίνει να προκαλούνται από πλειονότητα παραγόντων. Η μακρότερη καθυστέρηση που έχουμε σημειώσει είναι πέντε μηνών. Κι όμω ακούω τώρα για λογαριασμού που δεν έχουν πληρωθεί 1,5 χρόνο. Γιατί? Γιατί είναι πολύ περίπλοκες οι διαδικασίε μεταφορά, Δηλαδή από τη στιγμή που θα λάβουμε την αίτηση, θα την εγκρίνουμε κτλ. θα πρέπει να πάει από τα διάφορα επίπεδα, δηλαδή από το ευρωπαϊκό στο εθνικό, στο περιφερειακό μέχρι το τελευταίο δικαιούχο. πολλέ μεταφορέ ε, λοιπόν των κονδυλίων των πιστώσεων αυτών. Δική μα υποχρέωση συλλογικά είναι να εξετάσουμε τρόπους Απλούστευση των διαδικασιών αυτών. Κάτι που με ανησυχεί πολύ, πάρα πολύ, είναι ότι κάθε φορά που ξεκινά μια πρωτοβουλία απλούστευσης, αρχίζουμε μεν καλά, μετά η προσπάθεια αυτή περνά από πολλά επίπεδα διαβουλεύσεων, Συμβούλιο Υπουργών, Κοινοβούλιο, από τη στιγμή που είναι όλα πια έτοιμα, ίσως τα πράγματα να έχουν γίνει ακόμα πιο περίπλοκα αντί πιο απλά. Κάπου πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Από τη δική μου πλευρά σας βεβαιώνω ότι έχω την αποφασιστικότητα να απλουστεύσουμε. Ξεκινάμε από κάτι πιο περίπλοκο και καταλήγουμε σε κάτι απλούστο. Δεν πάνε το αντίθετο. Ομολογώ ότι προέρχομαι από ένα πολύ μεγάλο οργανισμό από την Παγκόσμια Τράπεζα και νόμιζα ότι ξέρω ότι θα πει γραφειοκρατία και τίποτε δεν μπορεί να με εκπλήξει. Αλλά έκανα λάθος. Διαπίστωσα ότι έχουμε περιττές περιπλοκές μέχρι σημείου που να μειώνουν την αξιοπιστία μας και να διαβρώνουν αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνης. Γίνονται όλο και πιο περίπλοκα τα πράγματα και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην προσπάθεια επιδίωξης αυτού του στόχου. Για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες χρειαζόμαστε μια διαδικασία που να εγγυάται την έκβαση, αλλά όχι παραπάνω βλέπουμε καμιά φορά το τέλειο να γίνεται εχθρό του καλού ή του καλύτερου. Στην Κομισιόν είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να διαρθρώσουμε διαδικασίες στην βάση του ότι must do, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει δουλειά χωρίς να το κάνουμε αυτό. Κάτι επίσης που μπορεί να είναι μια άλλη προσέγγιση να είναι ε, ενδεχομένω χρήσιμο αλλά όχι απαραίτητο. Αυτό πριν αναγκαίο πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Ελπίζω ότι θα μας χορηγήσετε την υποστήριξή σας έτσι ώστε να φτάσουμε. Αυτή η επιχρήσωση των κανόνων είναι ένα μαζικό πρόβλημα. Έχω δει αποφάσεις με 40 υπογραφές για μια έγκριση πληρωμής όταν θα είχαν αρκέσει 4 υπογραφές. Και μπορώ να σας πω ότι οι υπόλοιπε 36 υπογραφές δεν ευθύνεται για αυτές οι κομισιόν προέρχονται. Διακόπτει ο πρόεδρο. Μήπω επειδή είναι πάρα πολύ υπερβολικό το διοικητικό βάρο και ο καθένα ο καθένας θέλει να βάλει το χεράκι του μέσα. Να λοιπόν από πού προέρχεται όλη αυτή η περιπλοκότητα. Ναι, ναι, δε, η κυρία Γεωργίευα. Όταν ανακατεύονται, μάλλον όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο πειθαρχημένε. Ο πρόεδρο διακόπτει. Χωρί μικρόφωνο και λέει κάτι το, κάποιο αφιολόγημα. Δεύτερο λοιπόν, συνεχίζει η κυρία Γεωργίουδα θεωρώ ότι οι τελικοί δικαιούχοι, τελικά, αυτοί υφίστανται πρωτίστως τις αρνητικές συνέπειες. Γι' αυτό λέω ότι, και αυτό έχω τονίσει τόσο πολύ, αυτή την ανάγκη να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται να δημιουργηθεί, να εξεταστεί μάλλον πιο έντονα, είναι πού εντοπίζει το κίνδυνο, δηλαδή τι κινδυνεύουμε να χάσουμε εάν δεν εκτελέσουμε αποτελεσματικά τα προγράμματά μας. Άκουσα από διάφορους ομιλητές να δίνουν έμφαση ε, σε ξεκάθαρες προτεραιότητες, ξεκάθαρους στόχους και πολύ σημαντικό αυτό, να γίνουν αυτά τα πράγματα διαφανή για τους πολίτες, στα μάτια των πολιτών. Διότι ο καλύτερος έλεγχος, οικονομικά μιλώντας, είναι η διαφάνεια και η ανάληψη ευθύνη που προέρχεται από αυτήν, η λογοδοσία. Να ένα σημαντικό πρόβλημα που θα δούμε πώς θα το λύσουμε. Γιατί είμαστε βεβαίως πολύ διαφανείς, μάλιστα τόσο διαφανείς, τα δημοσιεύουμε, δημοσιεύουμε τα πάντα με τόση ε, εξαντλητική λεπτομέρεια, ώστε τόσο πολλά δέντρα κρύβουν τελικά το δάσος στα μάτια των ε, πολιτών. Δεν μπορείς να βρεις αυτό που ψάχνεις, διότι είναι χαμένο μέσα σε απίστευτες λεπτομέρειες. Μιλήσατε για αυτή την πολλαπλότητα των ελέγχων, για ε, έλεγχους και τήρηση ισορροπιών. Τελικά τα χάνουμε, χάνουμε τη λεπτομέρεια μέσα στο σύνολο αυτό των ρυθμίσεων. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς... Ναι, έχουμε βέβαια μακροοικονομικές απαιτήσεις. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαρες σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Αυτά όμως πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία με μια έμφαση στην ανάπτυξη και στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Για την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το συνέστημα κυριαρχεί. Είμαι βεβαία ότι το ακούσατε και από τον πρόεδρο Γιούνκερ και θα το ακούσετε και από τους άλλους και άλλες συναδέλφους μου. Τέλος, μια ερώτηση που ε, είχε το περιεχόμενο αν μπορούν να επιτευχθούν μέσα στο παρόν πλαίσιο μακροπρόθεσμοι λύσεις. Ναι, μπορούμε βέβαια να ισοσκελίσουμε τα βιβλία μας υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζουμε τους περιορισμούς που επιβάλλει το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναλάβουμε υπερβολικές δεσμεύσεις, πρέπει να είμαστε πιο ε, προσεκτικές. Βέβαια, τα, στα βιβλία μπορούμε να τα βρούμε, μπορούμε να τα ισοσκελίσουμε, αλλά δεν είναι εκεί το πραγματικό ερώτημα. Έχουμε τις σωστές προτεραιότητες και ο προπολογισμό μας είναι επαρκής για τις προτεραιότητες αυτές. Κάποιος είπε γιατί δεν φτιάχνετε μεγαλύτερα έργα, χρηματοδοτείτε μεγαλύτερα έργα και όχι μια πληθ, πληθώρα μικρών αν θέλετε να πετύχετε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Μα εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα μεγέθους. Μικρά έργα καμιά φορά έχουν ε, σημαντική κοινωνική απήχηση. Προσφέρουν πολλά. Τα ακούσατε αυτά ε, και από ορισμένου ομιλητέ σα. Συμβαδίζει ο στόχος και η πόροι Αυτό είναι το ερώτημα. Και μπορούμε να τα κάνουμε αυτά με επιτυχία με τον τρόπο που συγκεντρώνουμε τα χρήματα τώρα και 80% των πόρων της Ένωσης που έρχονται από εθνικές συνεισφορές μετά από πικρές και ε, δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να βελτιώσουμε και το διαπραγματευτικό περιβάλλον, να έχουμε ξεκάθαρους στόχους και ευθυγράμμιση επί των στόχων αυτών, με πολύ λιγότερο πικρό και διαιρετικό τρόπο από αυτόν που είδα στις πρώτες μου εμπειρίες ε, διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς δεν κατέληξαν επιτυχώς. Αν θέλουμε όμως να είμαστε επιτυχείς στο μέλλον πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους στόχους, να ευθυγραμμιστούμε με τους στόχους αυτές και τις προτεραιότητες μας και να είναι επιτυχής προσπάθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τώρα ε, για το χρόνο σας. Μήπως υπάρχουν και δικαστικές διαδικασίες λόγω των καθυστερημένων αυτών ε, ε, πληρωμών. Έχουν γίνει αγωγές κατά της Κομισιόν. Όχι, δεν γνωρίζω προς το παρόν μια τέτοια νομική υπόθεση, δικαστική υπόθεση εναντίον της Κομισιόν. Γνωρίζω ότι υπήρξαν ε, διαμφισβητήσεις σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με την πρόοδο των πληρωμών. Αλλά από ό,τι ξέρω δεν υπήρξε δικαστική ενέργεια κατά της Κομισιόν. Νομίζω ότι το επιβεβαιώνει και συναδελφοί μου. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουμε ακόμα μια τέτοια περίπτωση και ποιος ξέρει μήπως ε, όσο μιλάμε γίνεται κάτι. Το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μια τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να μας δίνει ρόλου ε, λόγω εφησυχασμό. Γιατί έχουμε ακόμα 25 δισεκατομμύρια τα οποία δεν έχουμε πληρώσει και μας δώστηκαν παραδείγματα του τι σημαίνει να μην πληρώνονται αυτά τα δισεκατομμύρια από αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο πριν από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ βασιζόμαστε σε εσά για να βελτιώσετε και να απλοποιήσετε τι διαδικασίε και τα κράτη-μέλη επίση πρέπει να κάνουν τι απαραίτητε προσπάθειε. Δεν είναι μόνο η οποία δημιουργεί πολυπλοκότητα. Πολλέ φορέ οι εθνικέ διοικήσει έχουν μια, ένα φετιχισμό με την πολυπλοκότητα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια πρόοδο κατά τα άλλα. Εμεί βασίζουμε πολλέ ελπίδε στην ε, αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου η ελπίδα μας είναι ότι δεν ήταν απλώς μία καινή δέσμευση που ελήφθη από το Συμβούλιο όταν έγινε η έγκριση του πλαισίου για να χρυσώσει το χάπι, αλλά θα είναι μια πραγματική υποχρέωση και επομένως θα είναι μια ουσιαστική ε, τροποποίηση, διότι η συμφωνία για το πλαίσιο έγινε πριν από τις ευρωεκλογέ. Ελπίζουμε ότι με την ευκαιρία αυτή τα κράτη-μέλη θα καταβάλουν μια προσπάθεια να επιληθεί το πρόβλημα των απλήρωτων λογαριασμών. Γιατί έχουμε φτάσει πια στα όρια του δυνατού και όπως τονίσατε και εσείς κυρία Επίτροπε είναι απόλυτα απαραίτητο να εξασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία που βρίσκεται σε κίνδυνο τώρα. Σας ευχαριστούμε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές. ο κύριος Σουντάν, ίσως έχω δολοφονήσει το όνομά σας βέβαια, Ζιρκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ωραία το είπατε το όνομά μου κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η κρίση πληρωμών οδηγεί και σε απώλεια αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των σχεδίων και η δυνατότητα να εφαρμοστούν σωστά τα σχέδια αυτά. Σίγουρα με την επερχόμενη μεταρρύθμιση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνεχής ενασχόλησή μας ώστε να μπορέσουμε να επιφέρουμε πιο εύκολα τις διορθώσεις όταν είναι απαραίτητο και να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στα μελλοντικά σχέδια δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια οριστική λύση γιατί αυτό σημαίνει να καταβληθούν όλα τα οφειλόμενα. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι θετικό είναι η χρήση των τραπεζών αναπτυξιακού χαρακτήρα στα κράτη-μέλη. Να υπάρξει λοιπόν και μεγαλύτερη εμπλοκή τους στη διαδικασία εφαρμογής των σχεδίων αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα απαιτούνται τόκοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω καθυστέρησης. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις τράπεζες επενδύσεων των κρατών μελών ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να είμαστε πραγματικά λειτουργικοί, να έχουμε μια πιο γρήγορη χρηματοδότηση και να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς μας και την εξισορρόπησή τους και εδώ έχουμε ένα ακόμα στοιχείο το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε γιατί έχει πραγματική επίπτωση υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό θα είναι αποφασιστικό για τους μελλοντικούς μας προϋπολογισμούς. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κουατία Σαμπάλ που ήταν ε, η συγγήτρια το, για το 2015. Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν αποφασίσαμε στους συντονιστές να θέσουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, νομίζω ότι είχαμε δύο στόχους να το συζητήσουμε το θέμα με τα Εθνικά Κοινοβούλια, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της μη, των μη καταβολών και να το δούμε από πρώτο χέρι και νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία. Το είδαμε με τους τρεις προσκεκλημένους πώς δεν γίνονται αυτές οι καταβολές στις τοπικές αρχές και στις περιφέρειες και νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε την υποστήριξη των Εθνικών Κοινοβουλίων όπως ε, γνωρίζετε και ενώπιον της Επιτρόπου μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε στη διαπραγμάτευση των ε, προϋπολογισμών. Ήδη από το 10 υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και γνωρίσαμε και μέχρι τώρα αυτές τις δυσκολίες, μέχρι το 2015. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε ε, θεωρητικά του, τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο, αλλά στην πράξη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, πρόκειται για μια διαλκυστίνδα με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θέλει να επιβάλλει ε, τα δικά του και βεβαίως σε μας ε, έγκυται να αντισταθούμε. Δεν ξέρουμε κάθε φορά πώς το Κοινοβούλιο μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και γι' αυτό θα πρέπει οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει με την μη καταβολή πληρωμών, γιατί χρειάζεται να πιέσετε κι εσείς τις εθνικές κυβερνήσεις για να δεχτούν το ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι σημαντικός, αφορά επενδύσεις και πρέπει να γίνουν οι καταβολές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτά τα ελλείμματα τα οποία είναι και παράνομα. Δεν ε, μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο. Ε, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση δεν ε, πληρώνουμε και είναι το ίδιο σαν να πρόκειται για ένα έλλειμμα. Θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από τα Εθνικά Κοινοβούλια έτσι ώστε να πιέσουν τις κυβερνήσεις και στην Επιτροπή Οικονομικών ή στις μικτές επιτροπές να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός μας. Ως προς τις καθυστερήσεις της πληρωμές, κατά πόσο θα υπάρχουν χρηματικές ποινές ή όχι, κατά πόσο υπάρχουν τόκοι υπερημερίες και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, η έλλειψη περιμεριες και ουτω καθεξης δυστυχως γίνεται στην πολιτική συνοχή, δηλαδή Εκεί που χρειάζονται περισσότερο οι πληρωμές, δυστυχώς εκεί βλέπουμε ότι πλήττεται περισσότερο ο τομέας. Και αυτό αφορά τα ίδια τα κράτη-μέλη, δηλαδή προκαλούνται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό δεν γίνεται και καμία καταγγελία, γιατί δεν μπορεί ένα κράτος να αυτοκαταγγελθεί για μη καταβολή. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι από μία πλευρά λέμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει την οικονομική της πολιτική. Θέτουμε μία πολιτική επενδύσεων, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο μέσο που έχουμε, το πρώτο επενδυτικό μέσο που είναι ο προϋπολογισμός μας. Συγχαρητήρια γιατί επιλέξατε αυτό το θέμα και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και να έχουμε την υποστήριξη των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπόρτς Βέσλουντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Απλώς γιατί θέλω να υποσχεθώ στους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο κάτι. Τα εθνικά μας κοινοβούλια δεν μπορούν όλα να σας βοηθήσουν, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να τεθούν σαφείς προτεραιότητες. Έχουμε διαφορετικούς στόχους, έχουμε διαφορετικό κόστος ο καθένας. Δεν είναι δυνατόν όλα τα κονδύλια να μπαίνουν στο, σε ένα τεράστιο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χωρίς να πληρώνουμε για την κοινωνική ασφάλιση, για την περίθαλψη. Δεν είναι δυνατόν να τα κάνουμε όλα συγχρόνως. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Γιατί, Γιατί πρέπει πραγματικά να τακτοποιηθεί η κατάσταση. Εμείς σε εθνικό επίπεδο μπορούμε ελάχιστα να επηρεάσουμε. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε οδηγίε στους υπουργού μας, αλλά ω εκεί, τίποτα περισσότερο. Συνεπώ αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει διάλογος. 15 χρόνια είμαι στο Ρίξταγκ και ποτέ δεν συμμετείχα σε κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει επιτέλους. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι με μεγάλα προγράμματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να φουσκώσουμε ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα ήταν λάθος κάτι τέτοιο και πολύ λάθος για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Δεν νομίζω ότι οι Σουηδοί εκλογής θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο από τα 2 δισεκατομμύρια κορώνες που εμφυσεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό η Σουηδία σήμερα. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κονδυλία στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτοί όμως που πληρώνουν είναι οι χώρες μέλη. Κανένας άλλος. Αυτό είναι σφάλμα για το όλο σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος αυτός, είναι αναγκαίος. Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Έχουμε εντελώ διαφορετικά σημεία κίνηση στις συζητήσεις που κάνουμε. Δεν πρόκειται μόνο για το φούσκωμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού, πρέπει να υπάρχουν και άλλα. Πολύ θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε να συζητάμε για, τα, για το με ποιο τρόπο θα βάλουμε τάξη στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δυστυχώς έφυγε η Επίτροπος. Τελικά ποτέ δεν εμπλεκόμαστε στις συζητήσεις. 15 χρόνια είμαι στο ρίξο στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα εκεί. Πρόεδρος. Άρα πρέπει να οργανώνουμε πιο συχνά τέτοιου είδου συνεδριάσει, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μα, να ανταλλάσσουμε απόψει, ώστε να γίνεται σαφέ το ότι απασχολεί το καθένα. Ο ρίκ Βαντερπόιερ έχει τώρα το λόγο. Είστε εδώ. Ναι, είμαι Φαν Ρομπάου, είμαι αδερφός του Προέδρου, του Χέρμαν Φαν Ρομπάου να μεταφέρετε τους χαιρετισμού μας στον πρόεδρο Φαν Ροπά, παρακαλώ. Βεβαίως, εγώ έχω μία ερώτηση. Αυτά που λέμε για τις οφειλές, τους απλήρωτους λογαριασμούς όσον αφορά τα προγράμματα συνοχής, 24 εκατομμύρια λέμε. Και τι διαφοροποίηση υπάρχει στις χώρες με 4 δισεκατομμύρια μάλλον για την Τσεχία, 24 για την Ισπανία, 7,3 για την Ιρλανδία, 2,7 δισεκατομμύρια για την Πολωνία, Πορτογαλία 7 εκατομμύρια. Συνεπώς η διαφοροποίηση είναι τεράστια που υπάρχει όσον αφορά τις χώρες μας. Οπότε ρωτάω, πώς γίνεται αυτό. Δεν είναι ευθύνη της Ευρώπης, είναι ευθύνη των χωρών μελών οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο τελικά ελείψει αξιόπιστων πρωτοβουλειών τους, ελείψει ελέγχων και από την Ευρώπη και από τις χώρες μέλη έχουμε φτάσει σε αυτές τις οφειλές. Οπότε γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διαφοροποίηση από τα 24 δισεκατομμύρια και βλέπουμε ότι άλλες χώρες δεν έχουν σχεδόν καμία οφειλή και άλλες τέσσερα. Υπάρχουν τρεις χώρες που έχουν ε, απλήρωτους λογαριασμούς πάνω από τέσσερα δις. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο μεγάλες ε, διαφορές και συμφωνώ με τον Γερμανό συνάδελφο που λέει ότι μήπως έτσι περιορίζονται τα προγράμματα. Τελικά μήπως χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός σαν εφαλτήριο για μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα. Μήπως μεγαλύτερα προγράμματα ενεργοποιούνται αντί για χιλιάδες ε, συγχρηματοδοτούμενα μικρά και μεσαία προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να επιζήσουν χωρίς αυτή τη στήριξη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Καρέλ Φίτλερ, ο τελευταίος μας ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω εν συντομία σε αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα μετά. Αναφέρθηκαν κάποιες αφιβολίες σε σχέση με τον τωρινό μηχανισμό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ακούμε σήμερα μας κάνει ακόμα πιο ε, σίγουρος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι λύση το να περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα πρέπει να υπάρξει απλοποίηση των μηχανισμών, όπω είπαν και πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές. Νομίζω κάποιος ανέφερε προηγουμένως ότι, ότι θα πρέπει να πιο ρεαλιστικές οι απαιτήσει. Και έχω το εξής ερώτημα να θέσω. Η κυρία Γιώργεβα μας ανέφερε ότι οι κανόνες θα πρέπει να τύχουν απλοποίησης και να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Υπάρχουν πράγματι κάποια σχέδια να εξασφαλιστεί αυτή η απλοποίηση των κανόνων. Και πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, πότε μπορούμε να περιμένουμε να λάβει χώρα κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για την ε, παρέμβαση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλα αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι συνεδριάσεις. Νομίζω ότι αυτή η, διακυβεν... αυτή συγγνώμη, διάσκεψη, στην οποία εγώ έχω συμμετάσχει στο παρελθόν ως εκπρόσωπος της Γαλλικής Γερουσίας, στο παρελθόν με έφεραν σε κάποια μηχανία γιατί γύριζε στο Παρίσι από τις Βρυξέλλες, ρωτούσα τι ακριβώς είχα παρακολουθήσει, δεν υπήρχαν ούτε ημερήσεις διάταξης, ούτε πρόγραμμα, ούτε τελική ψηφοφορία και πάντα θεωρούσα ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πιο στενή σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια πιο συνεχή ανταλλαγή απόψεων. Όχι να υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μακριά στον οριζόντα τα Εθνικά Κοινοβούλια, χρειάζεται να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μα και να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που ετέθησαν. Και τώρα είναι ο ο ρόλος των συντονιστών που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε κάθε μία από τις, από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα των μη καταβεβλημένων οφειλωμένων ποσών, των ΡΑΛ. Υπάρχει πάντα αυτό το χάσμα μεταξύ πιστώσεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών. Και είχαμε ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια σε τέτοιες ε, πληρωμές. Υπήρχε λοιπόν ένα συνολικό, μια συνολική θέση 220 δισεκατομμύριων, πάνω από 150% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο τέλος του 2013, λέει ο πρόεδρος. Με συμφωνία λοιπόν μεταξύ των δύο σκελών της αρχής του προϋπολογισμού, το Συμβούλιο που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Εκεί βρίσκεται η πολιτική πράξη η σύναψη υποχρέωσης, ενώ η πληρωμή είναι απλώς η εκτέλεση μιας πολιτικής απόφασης εκεί. Χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια για να ασκηθεί πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και την υλοποίησή του. Καταλαβαίνω το μήνυμά σας που είναι να υπάρξει μια απλοποίηση και να εστιάσουμε τις προσπαθίες μας σε συγκεκριμένα σημεία. Αλλά το πολιτές πλαίσιο εφέτος ακόμα δεν μας επιτρέπει μια τέτοια προσαρμογή. Μήπως θα υπάρξει κάποτε κάποια λογική να μπορούμε να πάρουμε μακροχρόνιες υποχρεώσεις για τη συνεκτικότητα, τη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών μας. Για τα κάτι μελη μας αυτό είναι λογικό. Αλλά ένας ε, προϋπολογισμός που δεσμεύεται με 7 χρόνια πριν, αυτό δεν επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές στην πραγματικότητα. Εξού και η ανάγκη να συζητήσουμε καλύτερα τη λογική του πολιετούς πλαισίου που είναι τόσο μακροχρόνιο, που ουσιαστικά περιορίζει τον προϋπολογισμό, το βάζει σε ράγες που πολλές φορές δεν μας πηγαίνουν πουθενά. Κατανοώ αυτά που έλεγχαν για την απλοποίηση. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Και κάπου η δημιουργία θέσεων εργασία, θέσεων εργασία εθνικέ διοικήσει είναι κάτι το ευχάριστο για τι εθνικέ διοικήσει. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Σίγουρα χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι για να αποτρέψουμε ενδεχόμενες καταχρήσεις, αλλά συμφωνήσουμε για κάποιο είδος ελέγχου, να λύνουμε ποιος θα πρέπει να φέρει σε πέρα τον έλεγχο αυτό και θα πρέπει να είναι απλοί οι κανόνες. Οι πιο πολύπλοκοι, πολύ πιο πολύπλοκοι κανονισμοί είναι αυτοί οι οποίοι παρακάμπτονται πιο εύκολα και γίνεται εκεί πέρα και η δυνατότητα λαθροχειριών σε δημοσιονομικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε μεγαλύτερη απλοποίηση. Δυστυχώ έφυγε η κυρία Γιώργεβα πριν από το τέλος της συζήτησης. Κρίμα που δεν μπορούσε να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα. Ιδίω του κυρίου Φαν Ρομπάι σε σχέση με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μια χώρα μπορεί να παίρνει γρήγορες πληρωμές, ενώ άλλες χώρες περιμένουν και περιμένουν για σημαντικά ποσά. Θα διαβιβάσω το ερώτημα αυτό στην κυρία Επίτροπο και θα επανέλθω κύριε Φανερόμπεϊ με την απάντηση που θα μου δοθεί. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε από κοινού και για το θέμα του προσδιορισμού της προσθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι χρήσιμα, έχουν μια αποφασιστική σημασία σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μήπως περιέχουν και δαπάνες που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για μας. Το λέω αυτό στο φως των συμπερασμάτων του ελεκτικού συνεδρίου. Το θέμα δεν είναι να δαπανώμε είναι να δαπανούμε με χρήσιμο τρόπο στην ίδια μου τη χώρα. Βλέπω ότι ορισμένα εγχειρήματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καμία αποφασιστική σημασία για την απασχόληση και την ανάκαμψη. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα. Θα έχουμε ένα σεμινάριο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών όσον ούπο, όπου θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά μέσα στην Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει αυτό. Θα ήθελα τώρα να κλείσω. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τις ε, παρατήρησει και τις ε, παρεμβάσει σα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις μαρτυρίες που καταθέσατε, οι οποίες μας παρουσιάζουν και την πραγματικότητα του φαινομένου αυτού που μας απασχολεί πολλές φορές Υπάρχει και κάποια απόσταση μεταξύ των Βρυξελών και του Στρασβούργου και των επιτοπίων πραγματο, πραγματικότητων. Αν θέλουμε οι ευρωεκλογέ να έχουν διαφορετικό χαρακτήρα από αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν και να ξεπεράσουμε το υψηλό επίπεδο αποχής και το υψηλό επίπεδο απόρριψης της Ευρώπης και του ευρωσκεπτικισμού θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τη σχέση μας να την κάνουμε πιο ζωντανή <clears throat> τη σχέση μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι και τα θέματα του προπολογισμού μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε όλα αυτά. Θα ακολουθήσει ένα κοκτέιλ στον χώρο Γεχούντι Μενουχίν, στο πρώτο όροφο, όπως βγαίνετε δύο πατώματα κάτω, κατεβαίνετε τη σκάλα, πηγαίνετε στον πρώτο όροφο και εκεί στο χώρο για χούντι Μενουχίν θα σας αναμένει ένα κοκτέιλ. Το απόγευμα έχουμε την Σύνοδο Ολομέλειας στις 3 ε, παρατέτατο και σας ε, εύχομαι καλή διακοπή.